Ε, good evening. Good evening. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και σας βλέπω γεμάτους ενέργεια. Από το θόρυβο της αίθουσας το καταλαβαίνω. Δεν ακούει κανείς κανέναν από το θόρυβο. Ας ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες μας. Έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας στην αίθουσα αυτή. Ξέρω ότι τελείωσαν οι διακοπές και ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη δουλειά μας. Καταρχήν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνώ στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταρχήν όσον αφορά τη διερμηνία. Δεν έχουμε βουλγαρικά και ρουμανικά σήμερα. Δεν έχετε διερμηνία στα βουλγαρικά και ρουμανικά. Και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σας ζητώ συγγνώμη. Νιώθω άσχημα. Αλλά μετά τις διακοπές καταλαβαίνετε μπορούμε να το αποδεχτούμε. Λοιπόν, Άλλη ανακοίνωση του Προέδρου για την Ψηφιακή Ένωση. Η τέταρτη συνεδρία τη Ομάδα Εργασία θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στι Βρυξέλλε, 2 με 4 το απόγευμα, 2 ώρε. 2 με 4 λοιπόν το απόγευμα, 23 Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα καλύπτει όλα τα ζητήματα από την προστασία ευαίσθητων δεδομένων μέχρι την προστασία υποδομών. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μας είναι προσκεκλημένα και η βοηθή σας και η συμβουλή σας παρακαλώ να είστε παρόντες σε αυτή την τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ψηφιακή Ένωση. Τέταρτο σημείο, έγκριση των πρακτικών τα οποία έχετε στο φακελό σας. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 15-16 Ιουνίου. 2015. Αγαπητοί φίλοι, εδώ στην πρώτη γραμμή νομίζω ότι ακόμη σας ακούω να μιλάτε. Και τα πρακτικά της 23ης Ιουνίου, δύο συνεδριάσεις. πρακτικά των δύο συνεδριάσεων, αν δεν έχουμε σχόλια, εγκρίνονται τα πρακτικά. Δεν έχουμε σχόλια. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε τις κάρτες μας όλοι. Βάλτε τις κάρτες σας λοιπόν. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Το ερώτημα της ψηφοφορίας είναι αν είστε χαρούμενοι που ξαναγυρίσετε στο κοινοβούλιο. Παρακαλώ απαντήστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Βλέπω έναν παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Πατρίτσια. Πέρασε της ψηφοφορίας. Α, βλέπω μεγάλη ευτυχία που ξαναγυρίσαμε. Χαίρομαι που η ψηφοφορία είναι ευτυχής που ξαναρχίσαμε τη δουλειά μας. Είχαμε και κάτι αποχές βέβαια. Να αρχίσουμε τώρα με την ψηφοφορία. Θα διαβάζω μόνο τα δύο τελευταία νούμερα των τροπολογιών. Καταρχήν 5228 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2-9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 8 0508 εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 00 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 01 υπέρ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 04 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 06 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για τη 06 ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 06 ψήφισαν όλοι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 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 05 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 06 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 07 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 0,8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 0,9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά. Να το ξαναπώ γιατί έκανα λάθος και είπα εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 05 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 Κύριε Μπουτικόφερ, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 04 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, Θέλετε να ελέγξουμε τη 13 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία. Για τη 13 λοιπόν, έλεγχος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Έχουμε έναν παραπάνω από τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 00 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 01 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 02 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 03 υπέρ, κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο. Για την τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ πολύ. 61 Συνολικά 50 υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε τον εισηγητή και περνάμε στο επόμενο σημείο. Τελική ψηφοφορία. Και το θέμα είναι για μια νέα συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι, COP21. Θα δούμε τις, τις τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες. Ένα υπέρ, κατά, αποχές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά επαλήθευση για το αποτέλεσμα για την τροπολογία 11. Ένας επιπλέον από τους σοσιαλδημοκράτες, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 ωραία επαλήθευση της 7 ψήφισαν όλοι Ένα επιπλέον από τους δεσσελιαλιστές, συγγνώμη πέρας τη ψηφοφορίας απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 σε δύο τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, επαλήθευση για τη 14 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της 14. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε και εδώ επαλήθευση δεν είναι σαφές άρχεται η ψηφοφορία και πάλι έχουμε έναν επιπλέον από τους σοσιαδημοκράτες πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό 17 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 17 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε μια παλήθευση και πάλι άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε και πάλι άρχεται η ψηφοφορία 21 Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας, παρακαλώ. Πρέπει να το απαληθεύσουμε γιατί δεν βλέπω τι θέλετε. 25. Επαλήθευση της 25. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά πρέπει να το επαληθεύσουμε και πάλι την 31 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 υπέρ κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε και πάλι. Για την 32 άρχεται η ψηφοφορία και τώρα πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές. Συγγνώμη πάλι πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 33. Πέρασε της ψηφοφορίας Πάλι έχουμε έναν επιπλέον από τους σοσιαλδημοκράτες. Πέρα της ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές να το επαληθέσουμε 45 πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές να την επαληθέσουμε και αυτή 47. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές έκρινεται, 55 υπέρ. Κατά να επαληθεύσουμε την 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές. Να το επαληθεύσουμε. 59. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μια μικρή διαφορά. 61 υπέρ κατά αποχές δεν καταλαβαίνω. Θα ήθελα να παρακαλέσω το ΕΛΚ να ψηφίζει λίγο πιο ξεκάθαρα. Επαλήθεση για το 61. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές 69 να κάνουμε μια επαλήθευση δεν είναι σαφής και πάλι συγγνώμη 69 πέραση της ψηφοφορίας Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές να το παληθεύσουμε 73 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορία εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Πάλι. Ζητώ συγγνώμη, 80. Άρχεται η ψηφοφορία για την 80 πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά απόχε εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι καταλαβαίνω. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 99 υπέρ, κατά αποχές, να την επαληθεύσουμε. 99. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθέσουμε και πάλι. Συγγνώμη. 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Βλέπετε. Έπρεπε να γίνει ο έλεγχος. 104 υπέρ. Προφορική, έχει προφορική τροπολογία από τους σοσιαλδημοκράτες Υπάρχουν ενστάσεις. Βάσει κανόνων θα πρέπει τουλάχιστον τέσσερα μέρη. Παρακαλώ σηκωθείτε, όπως στην Ολομέλεια. Υπάρχουν ενστάσεις, ε, αρκεί νομίζω, πάνω από τέσσερις. Ε, αυτό προβλέπει ο κανονισμός, ε, ζητώ συγγνώμη, όπως και στην Ολομέλεια. Ε, πρόκειται για τον κανονισμό, στην Ολομέλεια θέλουμε 39 άτομα, στην Επιτροπή χρειαζόμαστε 4 μέλη. Αυτό έχουμε αποφασίσει βάσει κανονισμού. Άρα ψηφίζουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. 104 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά μπορούμε και να το επαληθεύσουμε αν θέλετε. Ωραία, να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε, αλλά μάλλον εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Για την 105 εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίζεται 5 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 3 υπέρ κατά. Να επαληθεύσουμε το τρίτο τμήμα της 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το τελικό αποτέλεσμα για απόψε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εισηγητές μας. Η ψηφοφορία ήταν πολύ ομαλή, ένα διαδικαστικό. Μια Σύντομη παρατήρηση παρόλο πολύ θέλουμε να τελειώσουμε. Να ευχαριστήσω τον ασχετή τον κύριο Κέλλη που με τον οποίο είχαμε άριστη συνεργασία, νομίζω ότι οι ομάδε, όλε οι πολιτικέ ομάδε προτίμησαν τη δουλειά σα. Απλώ αυτό που είναι σημαντικό και θέλω να υποθεί είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε εδώ πλειοψηφία. Στην Επιτροπή μας φάνηκε ότι είχαμε βρει πλειοψηφία χάρη στην ηγεσία του κυρίου Κέλλη. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε στη σωστή πορεία. Μάικρο. Thank you very much. Rapporteurs and shadow rapporteurs. Oh. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και τους πιο εισηγητές. Πάμε στο επόμενο σημείο στην εμμυρίσή διάταξη. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Φίλοι μου. Well, we could... Μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε 35 λεπτά. Θα ήταν πολύ ωραία, αλλά παρακαλώ να ξεκινήσουμε αμέσω. Μια βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία για τα, για τα βασικά μέταλλα. Πολύ σημαντικό. Εισηγητή ο Εντουάρ Μαρτά. Να σα θυμίσω, συναδελφοί, ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών εξέπνευσε στι 10 Ιουλίου 2015. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, συνάδελφοι, εσεί στο διάδρομο, σα παρακαλώ, Φύγετε αμέσω από την αίθουσα, αφού δεν θέλετε να μας ακούτε. Παρακαλώ μη φιλιάστε δημοσίως. Αγαπητοί φίλοι από τους πρασίνους. Πράσινοι έξω και μέσα. Δεν μ' ακούνε καν. Ο συνάδελφο λοιπόν εντό ήταν με πολύ σημαντική έκθεση, με προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που εξέπνευσε στι 10 Ιουλίου 2015. Με 218 τροπολογίε ω τώρα. Έχουμε προβλέψει μια ώρα για τη συζήτηση και να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μαρτά. Έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά. Επίτηδε το κάνετε. Κάθε φορά μου στερείτε χρόνο. Έχετε κάτι εναντίον μου κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος διότι είναι αργά και ε, δεν είναι πολύ σύνηθες να έχουμε τέτοια ώρα τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε τόσο καλά όσο ο κύριος Κέλλη αρκεί να μείνουν όλοι και να ακούσουν τη συζήτηση στο τέλος. Απλώς ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε 280 τροπολογίες ε, και ότι το σύνολο των πολιτικών ομάδων και όλοι οι βουλευτέ δίνουν μεγάλη σημασία στο μέλλον τη ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίω σε αυτό τη βιομηχανία βασικών μετάλλων. Κοιτάζοντα το σύνολο των τροπολογιών, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενε απόψει ή μεγάλε βαθιέ διαφωνίε Λίγο πολύ συμμεριζόμαστε τις ίδιες ε, διαπιστώσεις. Υπάρχουν ε, τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία στα οποία συμφωνούμε όλοι. Πρώτον, η σημασία των βαστομετάλλων για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους τους ε, τομείς που αξιοποιούν αυτά τα μέταλλα, όπως η αιωλική ενέργεια, η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία και επίσης ότι η αναβιομηχάνηση της Ευρώπης περνάει από τα βασικά μέταλλα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τα βασικά μέταλλα ε, και ότι εδώ ε, η τιμή του άνθρακα που απειλείται με τις δωρεάν ποσοστώσεις και την ενδεχόμενη αύξηση του άνθρακα και επίσης τα μέτρα κατά του dumping διότι δεν μπορεί να είναι τελείω ανεξέλεγκτο ο ανταγωνισμό. Αυτά είναι δύο σημαντικά σημεία. Και τρίτο ε, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η διακύμανση των τιμών, ε, ιδίω τη ηλεκτρική ενέργεια, που οδηγεί σε από επένδυση στον ε, τομέα αυτό. Επί τη ουσία τώρα, νομίζω ότι ένα από τα βασικά μέτρα που προτείνουμε τον έλεγχο στα σύνορα δεν είναι κάτι που αντίκειται στην, ε, στο νέο σύστημα ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εκπομπών, ακόμη και όταν αυτό αναθεωρηθεί, αλλά πρέπει να προωθήσουμε τι επενδύσει χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, κάτι που έχουν στηρίξει το σύνολο των μηχανών που έχουμε συναντήσει ανά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό θα τους ε, ε, ευνοήσει αυτούς που προωθούν τα συστήματα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα σε σχέση με τους βασικούς τους ανταγωνιστές. Εάν λοιπόν θέλουμε ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιμηχανία, προ όσου ασχολούνται και ενεργοποιούνται εκεί, για να έχουμε τι απαραίτητε επενδύσει. Να φανεί δηλαδή ότι ανταμείγουμε αυτούς που ε, σέβονται τους κανόνες ε, και όχι αυτούς που δεν τους σέβονται. Οι κανόνες ε, οφείλουν να γίνονται σεβαστοί από όλους. Και αυτοί που ακόμη αμφιβάλλουν για τις διάφορες δυνατότητες, να θυμίσω εδώ την οδηγία REACH ως παράδειγμα για την αξιολόγηση, αξιοποίηση μάλλον των τεχνικών γνωσιών μας, κανείς δεν την έχει αμφισβητήσει, όλοι την χαιρετίζουν. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία λοιπόν που παρομοίω πρέπει να ακολουθήσουμε στο ίδιο πνεύμα με την προσαρμογή στα σύνορα, κάτι που είναι ένα μέτρο ε, Εάν τέτοιο μέτρο δεν, προληφθεί και, δεν προβλεφθεί και έχουμε προστατευτικά μέτρα, ε, θα έχουμε πίεση από ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα ε, με τον, ε, με τον ισότιμο ανταγωνισμό θέλουμε να ανταμείψουμε τους ε, παραγωγούς που σέβονται τους κανόνες για να γίνουν και απαραίτητε επενδύσει, όπω είπα προηγουμένω, υπέρ τη ενεργειακή αποδοτικότητα και των νέων τεχνολογιών, που θα μα επιτρέψουμε να εκπέμπουμε όσο λιγότερο διοξείδιο του γίνεται. Να θυμίσω επίση ότι με την έκθεση που ψηφίσαμε πρόσφατα, είδαμε ότι στο σύνολο των χωρών είδαμε πώς μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποστείλει ισχυρά ενήματα. Εδώ λοιπόν η προσαρμογή στα σύνορα είναι σημαντική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλλά και ως εργαλείο για να έχουμε την αναβιομηχάνηση ε, και να έχουμε και τις απαραίτητες επενδύσεις. Υπήρξαν κάποιες τροπολογίες, τις υποστηρίζω διότι μας επιτρέπουν να δούμε αυτό το μέτρο ως και ένα οικονομικό μέτρο για τους πράσινους στόχους μας. Έχουμε ούτως ή άλλως ε, την ανάγκη να βρούμε ένα κονδύλι 100 δις ε, δολαρίων για να ε, μπορέσουμε να στηρίξουμε τους δεσμευτικούς ελπίζω στόχους που θα αποφασιστούν στο Παρίσι σύντομα και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις μας η υποχρέωση πληροφόρησης και διαφάνειας. Βλέπουμε ότι σχεδόν όλοι οι βουλευτές ομόφωνα θέλουν τέτοια διαφανή πληροφόρηση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων από όλες τις πολιτικές ομάδες που μα στήριξαν ιδίω ω προ την πρόθεση των καλών πρακτικών για να περιοριστούν οι εκπομπέ του άνθρακα από τι βιομηχανίε βασικών μετάλλων και η δυνατότητα των οικονομικών και λογιστικών μέτρων για να μπορέσουν να καταγράφουν σε πρώτες πληροφορίες οι εκπρόσωποι των συντηρητικών οργανώσεων και των ε, πληθυσμών των κοινοτήτων που κατοικούν ε, κοντά στις βιομηχανίες είναι σημαντικά στοιχεία. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και επιτόπιες επιτροπές για την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Υπάρχει άλλο ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να βρούμε συμβαστικέ λύσει, τον εξυγχρονισμό των ε, μέσων ε, εμπορική άμυνα, για τα οποία υπάρχει γενική συνένεση, όμω εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προσαρμογέ για να διευθυνθούμε καλύτερα τη θέση μα και να κάνουμε τα σύνταξη ορισμένων τροπολογιών. Ιδίω ω προ την ανάγκη να διευκρινιστούν τα μέτρα που θα πρέπει να αναλυφθούν και τα οποία ακόμη βρίσκονται υπό συζήτηση. Και να, υπογραμμίσω ολοκληρώνοντα, αλλά σχεδόν ολοκλήρωσα κύριε Πρόεδρε, ότι ομόφωνα θέλουμε να υπάρξει προώθηση τη κυκλική οικονομία με την χρήση των ανακεκλωμένων μετάλλων, ακόμη και αν ε, ε, παραμερίσουμε εν μέρη την πρωτογενή παραγωγή. Εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε την τιμή του άνθρακα υπό το πρίσμα των ανακυκλωμένων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν του ΜΑΝ και του ΔΕ και την Τετάρτη το πρωί θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση, ω την Τετάρτη μάλλον, για να καταλήξουμε στις συμβαστικέ λύσει. αλλά επί τη ουσία δεν υπάρχουν ε, βασικέ διαφωνίε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρο, ευχαριστώ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σα ε, για τι εξηγήσει που να δώσατε. Και τώρα δύο ή τρία λεπτά για τους ή για τους συντονιστές. Κύριε Σαλήνη, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Όπως ε, διαπιστώσαμε την τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω την πολύ θετική εικόνα ε, που έχουμε για τη δουλειά που γίνεται, διότι οι γενικές κατευθύνσεις και οι πυλώνες τους οποίους ε, ε, στήριξε την έκθεσή του εισηγητής είναι στοιχεία με τα οποία έχουμε και εμείς σύμπνια Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια επανεκκίνηση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας ε, έχοντας στο επίκεντρο τη βιομηχανία και κυρίως τη βιομηχανία βασικών μετάλλων ε, εντός της ευρωπαϊκής μας βιομηχανίας. Προσέχοντας φυσικά και όλες τις απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να διακυβέσουν αυτή την ανάπτυξη ξεκινώντας από τον ενεργειακό τομέα. Στο ενεργειακό ζήτημα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε θέσει και στο εσωτερικό της ομάδας μου το θέμα της συνοριακής προσαρμογής ε, έχει κάποιες αντικρουόμενες θέσεις και νομίζω ότι το πιο λογικό θα ήταν να επιτρέψουμε στον εισηγητή να μας εξηγήσει ε, επακριβώς ε, τι προϋποθέτει αυτή η μεταρρύθμιση και η άποψή μου είναι ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχω πει και στις σχετικές συνεδριάσεις ότι υπάρχουν κάποια κρίσιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατάλληλα benchmarks τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών για να φτάσουμε σε αυτό το σύστημα της ενεργειακή προσαρμογής και επομένως θα πρέπει το ζήτημα αυτό ε, να έχει ολοκληρωθεί με την ε, ψηφοφορία πριν ξεκινήσει η όλη συζήτηση για την εμπορία εκπομπών. Αλλιώς ε, δεν θα είναι δυνατόν να έχουμε σωστή εργασία. Όσον αφορά το άμεσο κόστος, ο εισηγητής πολύ σωστά επισημαίνει ότι το ε, γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι αποζημίωσης στην Ευρώπη δημιουργεί στρέβλωση στην αγορά. Επομένως, η κατάλληλη ίσως λύση θα ήταν να μην υπάρχει αποζημίωση του άμεσου κόστους. Ε, καταλαβαίνω την ανησυχία για το θέμα του ανταγωνισμού εγώ έχω την εντύπωση ότι η λύση είναι το ακριβώ αντίθετο. Να πρέπει όλοι να αποζημιώνονται καταλήλω για το άμεσο κόστο. Ε, στη χώρα μου, για παράδειγμα, έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Ε, έχουμε κατηγορίε τι οποίες ε, προσφέρεται καταλήλω μέσω ενίσχυση ε, από το κράτο και υπάρχουν και χώρες όπως η δική μου που δεν το κάνουν αυτό και αυτό είναι εις βάρος μας κατά την άποψή μας. Η λύση λοιπόν για να υπάρχει ισορροπία στην αγορά κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπάρχει ε, με ομοιόμορφη αποζημίωση σε όλες τις περιπτώσεις σε γενικές γραμμές όμως είναι θετική η στάση μου. Ε, το έργο του εισηγητή είναι πολύ σημαντικό. Ε, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις εγκαταστάσεις ίσως και μέσω των κατάλληλων ταμείων για την ανάπτυξη και του ε, ταμείου στήριξης και την Τετάρτη θα δώσουμε και την υποστήριξή μας και την άποψή μας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε ο κύριος ε, και από πλευράς ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαχτά για την επιμονή του σχετικά με τη σημασία της βιομηχανίας ε, βασικών μετάλλων στην Ευρώπη και για τη θέση της βιομηχανίας αυτής ε, στον παγκόσμιο χώρο. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη βιομηχανία στο σύγχρονο πολύπλοκο περιβάλλον και διοικητικά πολύπλοκο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, συνθήκες σε κάθε χώρα χωριστά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά τονίζουμε τη σημασία της βιομηχανίας των βασικών μετάλλων στην Ευρώπη και ελπίζω ότι και οι επόμενες συζητήσεις μας θα είναι εξίσου επικοδομητικές. Ποια είναι τα προβλήματα αυτής της βιομηχανίας δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης. Εδώ η δική μας πολιτική ομάδα, το ECR, ακολουθεί μια διαφορετική θέση από τη δική σας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μεγαλύτερο διοικητικό φόρτος και περισσότερη έλεγχη θα βοηθήσουν αυτό τον ιδιαίτερα πολύπλοκο τομέα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μας δείχνει πόσο ανεπαρκές και πόσο πολύπλοκο είναι το σύστημα ε, ανταλλαγής εκπομπών, ε, δικαιωμάτων εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος. Το ξέρουμε όλοι. Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη βιομηχανία που συζητάμε είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πόσο δυσκίνητο είναι το σύστημα αυτό. Προσβλέπω λοιπόν στις μελλοντικέ μας συζητήσεις, γιατί τώρα πλέον έχει καταστεί προφανές ότι το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και ίσως πρέπει να αρχίσουμε να αναζητάμε διαφορετικά συστήματα, όπως σωστά είπε ο κ. Μαχτά. Πολλές εισαγωγές ε, είναι προνομιούχες διότι δεν επιβαρύνονται από αυτό το διοικητικό σύστημα το οποίο επιβαρύνει ευρωπαϊκές και μόνο εταιρείες. Βέβαια το σύστημα αυτό ε, ε, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικής συζήτηση αργότερα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ που τονίζετε τη σημασία αυτής της βιομηχανίας των βασικών μετάλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Άλντε και για Μίλναρ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς χαίρομαι που πρόλαβα. Έπειτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους για την ωστόρα δουλειά τους. Η έκθεση δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει όλες οι πολιτικές ομάδες για το θέμα. Με πάνω από 200, 279 ανθρωπολογίες είναι πάρα πολλές. Ε, είναι κατεπήγον να υπάρξουν βελτιώσει και αλλαγέ σε αυτό το τομέα. Αυτό δείχνει η εξέταση του θέματο. Και η βιομηχανία των βασικών μετάλλων στην Ευρώπη θέλουμε να γίνει ανταγωνιστική σε διεθνέ επίπεδο και πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Βλέπουμε από την έκθεση και τι τροπολογίε που υποβλήθηκαν ότι αντιμετωπίζουμε δύο βασικέ προκλήσει εδώ. Πρώτον, η ανάγκη να δράσουμε κατά των κλιματικών αλλαγών και έπειτα να βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά ως Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικότερες ευθύνες μας να ε, συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία που κάποιες φορές φαίνεται να μην συνάδουν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά και με την μείωση των ε, τιμών ενέργεια για προ τη βιομηχανία. Και βέβαια στο πλαίσιο συζήτηση άλλων ε, θεμάτων που μα αφορούν όπω οι διαπραγματεύσει για το TTIP και η Ενεργειακή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ε, θίγουν πολλέ τροπολογίε όπως η δική μου, είναι ότι πρέπει να έχουμε ισότιμού κανόνες για την βιομηχανία βασικών μετάλλων. Να τονίσω το εξή εδώ και να είναι σαφές, ότι έχουμε την διάσκεψη των μερών 21 στις αρχές Δεκεμβρίου στο Παρίσι και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο αυτής της σημαντικότητα τη διάσκεψης, ιδίω εάν μιλούμε για την προσαρμογή του άνθρακα στα σύνορα και τα υπόλοιπα μέτρα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο και εκτό Ευρώπη. Εδώ λοιπόν ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα για την έκθεση και σα ευχαριστώ πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ε, μάλλον της Γκούρη, κυρία Λόπε Περμερού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για την έκθεσή του και το έργο του και φυσικά και όλους όσους έχουν εργαστεί από αυτής της έκθεση. Ε, η ομάδα μου έχει υποβάλει τρεις τροπολογίες ε, που θέλει να ε, έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό δέσμευσης για τα ανακυκλώσιμα και να αυξήσουμε τα ανακυκλώσιμα που θα μπορούσαμε να παράξουμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για μεγαλύτερε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα καθορίσουν ένα σημαντικό κοινωνικό και περιφερειακό επίπεδο συνοχή ε, που είναι απαραίτητο στο βιομηχανικό επίπεδο. Επίση, θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Ε, στην Ισπανία υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική επιχείρηση, η Κογκάς, ε, η οποία εργάζεται στην έρευνα και στην καινοτομία για το θέμα αυτό και ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόοδος για το θέμα των εκπομπών και της μείωσης τους. Ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε πρακτικές dumping και ταυτόχρονα να υπάρχει απασχόληση ποιοτική. Θα θέλαμε επίσης να δούμε τι γίνεται με το θέμα της διαρθρωτικής ε, ε, διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του κόστους ώστε να μην υπάρχουν μόνο κάποια ιδιωτικά ολιγοπόλια. Ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα στοιχεία της ευελιξίας στα πλαίσια της ε, σύναψης ε, βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, κυρίως των διμερών συμβάσεων στην περίπτωση ε, των πολύ ενεργοβόρων επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο επενδύσεων. Ολοκληρώνοντας να πω ότι θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και ελπίζω να έχουμε τις, όσο το δυνατόν μεγαλύτερους συμβιβασμούς σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την βιομηχανία της Ευρώπης που κατέστρεψε πάρα πολλές θέσεις εργασίας και θα πρέπει να δημιουργηθούν ξανά νέες θέσεις εργασία σε ένα βιώσιμο φυσικά πλαίσιο. Ευχαριστώ εκ μέρους του EFTD, ο κύριος Μπορέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του, κυρίως διότι είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε επιτόπου η ομάδα μας ε, υποστηρίζει τη ρεαλιστική προσέγγιση του εισηγητή και κυρίως την πρόταση να χρησιμοποιήσουμε τη συνοριακή προσαρμογή για να μπορέσουμε να ευνοήσουμε την πιο ισότιμη ε, ε, δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ Ευρωπαίων και επιχειρηματιών εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις τα μειονεκτικά στοιχεία και να ευνοήσουμε τις επενδύσεις. θα μπορούσαμε ταυτόχρονα να εργαστούμε συμπληρωματικά και σε άλλους στόχους, ε, τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και ίσως και ένα φόρο ε, ε στην κατανάλωση άνθρακα. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το θέμα των εκπομπών σε εξωευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσε να είναι και αυτό κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη μας. Σε κάποιες από τις τροπολογίες μας αναφέρουμε και το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες άλλες καινοτόμες ε, στρατηγικές ε, για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών. Θα ήθελα να επισημάνω και το γεγονός ότι εμείς θα θέλαμε να συμπεριλάμβουμε και τους ε, τοπικούς πληθυσμούς και τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ολοκληρώνοντας να πω φυσικά ότι είμαι καθόλου διατεθειμένος να συνεργαστούμε για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας που έχουν δυσκολίες και εδώ σας λέω ότι είμαι πλήρως διατεθειμένος να συνεργαστώ και με τον εισηγητή φυσικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Και τώρα περνάμε στους υπολείπους. Η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Εντουάρα για την ε, έκθεση. Εδώ δεν μιλώ για να υπερασπιστώ τις τροπολογίες μου, αλλά ως βουλευτής που εκπροσωπώ μια περιοχή που έχει μια πολύ ισχυρή βιομηχανία ε, βασικών μετάλλων. Βιομηχανία η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πληθώρα προβλημάτων από κάθε προέλευση και νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ζωτική σημασία καθώς και η συγκυρία είναι πολύ επίκαιρη. Δεν θα υπάρξει αναβιομηχανία τη Ευρώπη αν δεν έχουμε τέτοια βιομηχανία βασικών μετάλλων. και πρέπει να έχουμε τέτοια πολιτικά μέτρα που να ε, στηρίζουν την ε, βιομηχανία αυτή συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετάλλων. Χρειαζόμαστε βιώσιμη οικονομία και επειδή μιλάμε πάρα πολύ συχνά για την αποθήκευση άνθρακα και τα σχετικά μέτρα στην Επιτροπή αυτή, να πω ότι στη δική μου την περιοχή ξεκίνησε το πρώτο κλάστερ για τα βασικά μέταλλα και την, ε, βιομηχανική, την, ε, τις βιομηχανίες χημικ, για το πρόγραμμα αυτό, για το σκοπό αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό και από την άποψη της καινοτομίας και πρέπει να στηρίξουμε και τροπολογίες ε, όπως της Μία Πάτρικ ε, 209 για την αναβιομηχάνηση και την περισσότερο οικολογική προσέγγιση της βιομηχανίας. Όσοι ε, ακολουθούν τους κανόνες θα πρέπει να παίρνουν και τις ανάλογες αμοιβέ και τα δελτία για τις σωστές εκπομπές τους. Και θέλουμε να αποφύγουμε τον τον ανταγωνισμό και το dumping. Γι' αυτό η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον εξυγχρονισμό των αμυντικών μέτρων στο εμπόριο είναι πολύ σημαντικά και αυτό ακριβώς ζητούν και οι βιομηχανικοί μας κλάδοι ανά την Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. κυρία Κουμπούλα Μάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να ξεκινούμε με ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι μεγάλη σημασία για τη χώρα που εγώ γνωρίζω καλύτερα ε, την Φινλανδία που εξαρτάται όχι μόνο από τα δασοκομεία αλλά και τη βιομηχανία βασικών μετάλλων στο Κοινοβούλιο ε, ε, στη συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας είδαμε ότι πραγματικά μα σοκάρει τι ανταγωνισμό υπάρχει με χώρα που θα μπορέσω να κατονομάσω, παρόλο που δεν είναι διπλωματικό αυτό, την Κίνα που ε, καταπατά όλα τα μέτρα θεμετού ανταγωνισμού. Είναι τελείω ε, αθέμητο αυτό ο ανταγωνισμό και πρέπει να το δούμε λοιπόν και από τη διεθνή σκοπιά. Ο δίκαιο ανταγωνισμό όμω εντό Ευρώπη είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να απασχολήσει. Γι' αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει, να προτείνει κάτι για τα έμεσα κόστη και τι σχετικέ προθεσμίε. Ε, θα πρέπει να δούμε αν έχουμε μια θέση σε αυτό το νέο κοινοβούλιο, διότι δεν με νοιάζει τι έκανε η προηγούμενη θητεία στο κοινοβούλιο, είμαστε τόσο πολύ καινούργοι. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο έχουμε μια κοινή αντίληψη σε αυτή την Επιτροπή για το τι πρέπει να ε, ε, κάνουμε για να υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά το τι γίνεται με τι κατευθυντήριε ε, γραμμέ για τι κρατικέ βοήθειε και το κατά πόσον διαφυλάσσεται η ισοτιμία του ανταγωνισμού για την βιομηχανία λοιπόν, μετάλλων στην Ευρώπη. Εκεί χρειάζεται δικαιοσύνη στον ανταγωνισμό και εκεί πρέπει να έχουμε γενικότερε και σωστότερε κατευθυντήριες γραμμέ για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ε, ο θεμετός ανταγωνισμός πρώτα πρέπει να ξεκινήσει στην Ευρώπη και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στην διάσκεψη για το κλιματικές αλλαγές στο Παρίσι και στις υπόλοιπες εμπορικές διαπραγματεύσεις μας σε διεθνές επίπεδο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα ο μιλητής, ο κύριος Λάγκια, από την, ο πρόεδρος της ΙΝΤΑ, Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι μόνο προσκεκλημένος μιλητής, αλλά είμαι και αναπληρωματικό μέλος. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλή η συζήτηση που γίνεται γιατί η χαλιβουργία είναι μια βασική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να την ενισχύσουμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα μέσα που διαθέτουμε μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών, μέσω έρευνας. Παρ' όλα αυτά έχω κάποια προβλήματα με την, τις προσαρμογές στα σύνορα. Δημιουργούμε ένα νέο γραφειοκρατικό ε, σύστημα. Θα έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να επιβαρύνονται με συγκεκριμένα τέλη δασμούς. Δημιουργούμε δηλαδή ένα νέο πολύπλοκο σύστημα. Δεύτερον, έχουμε όλο και περισσότερο, περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ, ε, που διακινούνται μεταξύ συνόρων. Έχουμε όλο και περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές ε, προϊόντων, ε, τις οποίες δεν θέλουμε να παρεμποδίζουμε και φοβούμε ότι και αυτές οι προσαρμογές στα σύνορα μπορεί να είναι αντίθετες ε, με τους ε, ε, κανόνες ελεύθερης διακίνησης ή ακόμη και με τους κανόνες του ΠΟΕ. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διενέξεων. Επίσης δίνουμε και ένα πολιτικό μήνυμα με αυτά τα οποία κάνουμε. Αν βάλουμε ε, κάποια τέλη προσαρμογή στα σύνορα στις εισαγωγές με την Ουκρανία ε, ρίνουμε ή αποθαρρύνουμε τις εισαγωγές ε, από αυτή τη χώρα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να δούμε αν τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία του εμπορίου μπορούν να εξελιχθούν. Προς το παρόν το Συμβούλιο μπλοκάρει τέτοιου είδους εργαλεία και αν εμείς σε κάποια χώρα για ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει dumping ε, σχετικά με το περιβάλλον, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Και θα πρέπει τότε να προσαρμόσουμε το επίπεδο των κυρώσεων ούτως ώστε να μην υπάρχει dumping ως στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάιε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, ξέρει ότι και εγώ θα ήθελα ε, να ασχοληθώ με μια τέτοια έκθεση γιατί το Duisburg ε, που είναι και η εκλογική μου περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό σημείο για την ε, χαλιβουργία στην Ευρώπη και θα ήθελα και εγώ να εμπλακώ με το θέμα αυτής της έκθεσης. Ο χάλιβας είναι μια, ένα βασικό προϊόν, είναι ένα προϊόν από το οποίο ξεκινά μια αλυσίδα πολλών άλλων προϊόντων και στο παρελθόν ε, είχαμε σημαντική βιομηχανία την οποία δεν χειριστήκαμε με την κατάλληλη προσοχή και μερικές φορές ε, η Επιτροπή ευθύνεται γιατί με την πολιτική της έχει απομονώσει κάποιους τομείς ε, ένα δρόμο ακολουθούν οι πολιτικοί, ένα άλλο δρόμο ακολουθούν ε, οι εμπορικές πολιτικές και εμείς ε, ως ε, ευρωβουλευτές θα πρέπει να χειριστούμε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με αυτή τη βιομηχανία. Ίσως τώρα με την Επιτροπή Juncker να μπορέσουμε να φέρουμε κάποια σχετική ισορροπία στον τομέα αυτό. Ο Μπέχ νομίζω ότι ήδη ανέφερε πολλά σημεία που θεωρώ και εγώ σημαντικά. Και όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις για την εμπορική πολιτική, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ε, μια σωστή εμπορική πολιτική στην Ευρώπη που να είναι σωστή και έναντι του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να μην ε, παραβιάζουμε διεθνείς συμφωνίες. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τη μέση οδό μεταξύ όλων αυτών. Και υπάρχει και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Και η Πέτρα νομίζω πολύ σωστά ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, γιατί μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού θα ε, απαγορεύει να έχουμε μια εταιρεία που θα είναι η πρώτη εταιρεία στην Χαλιβουργία. Μπορεί... Ε, μια φινλανδική εταιρεία να μπορούσε να γίνει η εταιρεία που θα είναι η ε, πρώτη εταιρεία διεθνώς και θα έφτανε αυτή η εταιρεία να έχει ε, δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο θα μπορούσε να είναι βιώσιμη μια εταιρεία αυτή στην Ευρώπη. Δυσκολεύουμε δηλαδή τη ζωή μιας τέτοιας εταιρείας βάζοντας ε, ε, παροπίδες και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη διεθνή κατάσταση του κλάδου. Εάν θέλουμε να προστατεύουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται διάφοροι κλάδοι διεθνώς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Και αν υπάρχει κάποιο σφάλιμα θα πρέπει ακόμη και στις συνθήκες να το αλλάξουμε με την επόμενη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, η κυρία Μαρία Τελοσφόρες Γκίτο. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που είπατε και όλο το όνομά μου. Ελάχιστοι το κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται απολύτως τις ανησυχίες ε, όλων όσων μίλησαν προηγουμένως ε, για την ασφάλεια για την ευρωπαϊκή οικονομία και ευχαριστούμε τον κύριο Μαρτά για την έκθεση αυτή η οποία είναι πολύ λογική και πληρέστατη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή συγκριθή στην τελική της εκδοχή θα αποτελέσει τροφή για σκέψη για τη συνεχιζόμενη συζήτηση και που γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους δύο συνομοθέτες ε, και τις μελλοντικές συζητήσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στις συζητήσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δεν θα επεκταθώ εδώ γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος χώρος, αλλά θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θεωρούσε ότι η συνοριακή προσαρμογή είναι τμήμα της εργαλειοθήκης της. Είναι κάτι το οποίο έχει κατά νου εδώ και αρκετά χρόνια, τα έχουμε λάβει υπόψη σε αρκετές αξιολογήσεις επιπτώσεων και το και η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή είναι ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι ένα ακόμα μέσο το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι παρενέργειες της ε, αποτελεσματικής ε, ε, κλιματικής πολιτικής θα μετριαστούν μέσω αυτών των μέτρων ε, βραχυπρόθεσμα όμως ε, στη νέα πρόθεση του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας εκπομπών και μακροπρόθεσμα στο διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών που θέλουμε να έχουμε μετά το Παρίσι είναι οι κατάλληλες ε, δράσεις που χρειάζονται για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τα αποτελέσματα. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ανέφερε κάποιο. Κάποιο αναφέρθηκε στι μακροπρόθεσμε συμβάσει και τα ενεργειακά ζητήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κλάδο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στου Ευρωβουλευτέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξελίξει μια δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια τη Ενεργειακή Ένωση και ε, το σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς ε, θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες και υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για αυτές τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Ε, θέλουμε λοιπόν και τη συνεισφορά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνει υπόψη τη και εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά την ανακύκλωση και την πρωτογενή παραγωγή, όπω ξέρετε θα υπάρξει μια δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και την ανακύκλωση σε δευτερόγενέ στάδιο, αλλά και την πρωτογενή παραγωγή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ο εισηγητή μα ο συνάδελφο Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές, η συζήτηση είναι πλούσια και συνολικά, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν έχουμε πρόβλημα στο να συμφωνήσουμε στις περισσότερες διαπιστώσεις, ακόμη και αν πρέπει κάποιες, κάποια συγκεκριμένα σημεία να τα ε, αποσαφηνίσουμε για να δώσουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Διότι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να υπάρξει αναβιομηχάνηση αυτή τη Επίρου που έχει αποβιομηχανιστεί εδώ και 30 χρόνια ιδιαίτερω. Και σε αυτό το τομέα το γνωρίζω πολύ καλά, διότι από αυτόν προέρχομαι. Εκεί χρειάζεται εναρμόνιση και θα ευχαριστήσω τον κύριο Σαρλίνη από το ΕΛΚ για τη δουλειά που έκαναν και για τις τροπολογίες τους. Θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει στο σύνταξη μια συμβαστικής λύσης για το κατά πόσον πρέπει ε, η βοήθεια για το έμεσο κόστο να ε, αλλάξει ή τουλάχιστον να εναρμονιστεί. Θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την έλεγχο στα σύνορα για το επιπλέον διοικητικό αθώς, για το κατά πόσο αυτό βοηθά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Επιτρέψτε μου να σας ε, εξηγήσω για ένα λεπτό κάποια πράγματα θεωρητικά. Έχω ασχοληθεί με τη χαλιβουργία εδώ και 30 χρόνια και για όσους ε, δεν το γνωρίζουν ή τουλάχιστον δεν έχουν σωστές ε, πληροφορίες ή δεν έχουν σωστές πληροφορίες από την τηλεόραση να πω ότι η παραγωγή του χάλιβα από το εργοστάσιο μέχρι τον πελάτη ε, σημαίνει ότι για να έχουμε ένα τόνο χάλιβα έχουμε τουλάχιστον 10 έως 30 φορές ε, περισσότερη ύλη από την τελική χρήση του άνθρακα, δηλαδή του χάλιβα. Δηλαδή σε κάθε στάδιο της μετατροπής έχει ε, σημειωθεί η ώρα της μετατροπής, το όνομα του ε, υπεύθυνου υπαλλήλου, οι ε, μετρολογικές συνθήκες ακόμα, δηλαδή ε, ένα δελτίο ταυτότητας που ακολουθεί το κάθε τελικό προϊόν για 30 χρόνια. Για τους λομπίστες λοιπόν και όσους λένε θα αυξηθεί το διοικητικό άχθος, είτε είναι κακόπιστοι είτε δεν έχουν δει ποτέ πώς γίνεται η παραγωγή ενός τόνου τέτοιου προϊόντος. Διότι αυτό το δελτίο ταυτότητας είναι η καλύτερη εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας για τον πελάτη. Ο καταναλωτή θέλει να ξέρει από ποιε συνθήκε παράχθηκε το προϊόν, πώ, γιατί, πού και όλα τα σχετικά. Είναι λοιπόν μία επιπλέον γραμμούλα παραπάνω που λέει ότι για να παραχθεί το τάδε ε, προϊόν χρειάστηκε τόση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Παίρνει 30 δευτερόλεπτα παραπάνω να προσθέσει κανεί αυτή την επιπλέον γραμμή. Κατά τα άλλα, αντί για τα γυαλιά έβαλα τα ακουστικά, τέλο πάντων. Ε, είμαι λίγο αναστατωμένο. Ε, κατά τα άλλα, να πω απλώς για την έκθεση αυτή και εδώ θέλω να ολοκληρώσω. Ε, μιλάμε για την ε, ανάγκη να υπάρξουν έρευνες και κοινοτομία, να ε, χρηματοδοτήσουμε την κατάρτιση και τις επενδύσεις σχετικά για να παραμείνει εύρωστη αυτή η βιομηχανία και να πω ότι κάποιες φορές η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία επενδύει στην ε, έρευνα και την κοινοτομία, αλλά μένουμε κάθε φορά στο κατόφλι, χωρίς να ανοίξουμε την πόρτα. Ένα παράδειγμα που έδωσε μια συνάδελφος, η Ελκογκάς, στην Ισπανία. Ε, μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, 100% χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια για να μειωθούν οι κομπές του άνθρακα και ε, πετυχαίνει. 99% λιγότερο, λιγότερες εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν ε, τα περαιτέρω στάδια της έρευνας αυτής για να δούμε πώς μπορούμε να ε, κατακατήσουμε τον άνθρακα και να τον αποθηκεύσουμε. Εκεί λοιπόν σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης βλέπουμε ότι δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχει και η ικανότητα να αποθηκεύσουν και τόσο το καλύτερο. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης για να δώσουμε και μια νέα ζωή στον άνθρακα. Και για να ολοκληρώσω, επειδή βλέπω πρόεδρε ότι είστε έτοιμο να μου κόψετε το μικρόφωνο και δεν μου αρέσει αυτό, με αγχώνει, ε, να ολοκληρώσω λέγοντα τι είναι η προσαρμογή του άνθρακα στα σύνορα. Κάθισα και το σκέφτηκα σε όλε τι συνεδριάσει που κάναμε, είδαμε ότι δεν ήταν σαφέ τελικά. Δεν είναι ένα φόρο στα σύνορα τη Ευρώπη. Ποια είναι η βασική ιδέα όταν έχουμε περάσει από τις 10 ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να περάσουμε, από τους 25 εκπροσώπους βιομηχανιών που τελικά συναντήσαμε, βλέπουμε ένα βασικό πρόβλημα να το αναφέρουν όλοι. Η ανταγωνιστικότητα αυτή σχετίζεται με αυτό που θέλουμε εμείς συνολικά, την αύξηση της τιμής του διευθυντή του άνθρακα και επιτάμε την ε, τιμή της ενέργειας, αλλά για την τιμή του άνθρακα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε επενδύσεις στην Ευρώπη και να μην φεύγουν ε, εκτός Ευρώπης. Ο κύριος Γέν που ήταν μαζί μου στην Γκέτσπουργκ είδε ότι η Dixon Group Η Thyssen δεν θέλει να επεν... Ε, ο δεν θέλει επενδύσει πλέον εντός της Ευρώπης αλλά εκτός. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι θα πρέπει να επιτρέψουν στους βιομηχάνου να περάσουν στις επενδύσεις που θέλουν χωρίς να επεβαρύνουν το κρατικό χαρτοφυλάκιο με την απαραίτητη δικαιοσύνη και τον ισότιμο ανταγωνισμό που θέλουμε ε, για τους βιομηχάνους εντός και εκτός Ευρωζώνης. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε μια προοπτική για το μέλλον και εδώ θα ολοκληρώσω. Ε, πρέπει να δώσουμε μια προοπτική για το μέλλον για τους βιομηχάνους και τους επενδυτές ώστε να επενδύσουν εντός Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικολογίες ε, στις οποίες δεν θα με βρείτε σύμφωνο διότι το βασικό στοιχείο είναι να δώσουμε ε, ελπίδα στους ε, μηχανούς και να ανοίξει η πόρτα της αναμηχάνησης για την Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, βλέπω ότι ήταν συναρπαστική ομιλία σας διότι πραγματικά κατέχετε το θέμα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό, φανταστικό για το τέλος της συνεδρίασής μας. Η ολοκλήρωσή της άλλωστε εξαρτάται το μόνο από εσά. Θα μπορούσατε να μιλήσετε άλλα 15 λεπτά. Θα είχαμε μείνει εδώ περισσότερο. Διάφορα, κάτι να πείτε στα διάφορα, όχι. Επόμενη συνεδρίαση, 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και 22 Σεπτεμβρίου το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγες μέρες. That's okay.